του άρθρου 78 ε, του κανονισμού έχω υπογράψει, θα υπογράψω μάλλον με τον πρόεδρο του Συμβουλίου μία ε, απόφαση για μακροοικονομική υποστήριξη προς την Ουκρανία. Ερχόμαστε τώρα στα θέματα της σημερινή συνεδρίασης Ολομέλειας. Υπάρχει μία αίτηση διαδικαστικής παρέμβασης του κύριου Κόρβετ. Κύριε Κόρβετ, έχετε το λόγο.